Ξεκινάμε αγαπητοί συνάδελφοι τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήλθατε όλοι και όλες. Μετά από αίτηση του συναδέλφου μας του κυρίου Ταμπάτζη, προτείνω να προσθέσουμε στη μέση διάταξη την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα ε, προϊόντα, επεξεργασία προϊόντων καπνού και εμπορία του καθώ και συναφών προϊόντων στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με αυτή την τροποποίηση. Αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Αμέσως όμως. Αμέσως. Αμέσως. Έχω να σας, την χαρά να σας πω ότι η διερμηνία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να σας πληροφορήσω ότι η Μαρία Ζάιφιτσμπέργκερ, που η Μαρία, ναι, που έχει εργαστεί στην Επιτροπή μας για 15 χρόνια ως συνεργάτησα και θα πάει σε μια νέα θέση ως ε, διοικητικός υπάλληλος ε, για τα ανθρώπινα διαχείριση προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Διερμηνία. Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια για την ε, Επιτροπή μα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε μαζί μου να πούμε ότι η Μαρία ήταν πραγματικά η σπονδυλική στήλη τη Επιτροπή, Το κέντρο τη οργάνωση που ανταποκρινόταν σε όλε τις αιτήσει των βουλευτών. Ξέρουμε, ξέραμε ότι πάντα μπορούσαμε να βασιζόμαστε στην βοήθειά της και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα η Μαρία πάντα μπορούσε να βρει μια λύση. Νομίζω λοιπόν ότι εξ ονόματο όλων των συναδέλφων τη Επιτροπή Γεωργία θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Μαρία για τη θαυμάσια εργασία που έχει φέρει σε πέρα για την Επιτροπή Γεωργία και φυσικά να τη ευχηθώ την καλύτερη επιτυχία στα νέα τη καθήκοντα. Ευχαριστούμε και πάλι Μαρία και σχετικά θέλω να σας πληροφορήσω ότι η κυρία Σιντόνια Φοκαράση, η οποία ήδη εργάζεται στη γραμματεία μας, θα αναλάβει τις αρμοδιότητες της Μαρίας. Και μια δεύτερη συνεργάτης θα έρθει μέχρι το τέλος του χρόνου στη γραμματεία μας. Καλώς ήλθες λοιπόν Σιδονία και καλή τύχη στην εργασία σου. Πάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών συνεδρίας 20-21 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν ε, <clears throat> αντιρρήσεις μέχρι το τέλο τη συνεδρίασης, θα θεωρηθούν τα πρακτικά αυτά ότι έχουν εγκριθεί. Και πάμε τώρα στο σημείο 4. Ναι, έχετε το λόγο κύριε Βασιλόσκη. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ως Επιτροπή Γεωργίας θα ήθελα να ευχηθούμε περαστικά στο συνάδελφό μας κύριο Παπαστάμκο και να ευχηθούμε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό κοντά μας. Ευχαριστώ Αλμπέρτ. Φυσικά, φυσικά και εμείς ευχόμαστε ακριβώς το ίδιο. Σημείο 4. Ο κύριος Βατσεβόφσκι δεν έχει φτάσει ακόμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε παρόλα αυτά την ψηφοφορία χωρίς αυτόν. Έκθεση Βοτσεκόφσκι για την αντιμετώπιση της ε, απάτης και προστασία των, χρηματο... των δημοσιονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρμόδια επιτροπή για τα θέματα αυτά είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Λαμβάνω υπόψη ότι η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει μία μείωση των ε, ατασταλιών και επίσης μία μικρή αύξηση των ε, ποσών που εμπλέκονται. Ήταν 1.230 περιπτώσεις ε, ατυπίες οι οποίες παρουσιάστηκαν. Είναι 35% λιγότερο από το προηγούμενο έτος. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν να κάνουν με την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και να υπάρξει καλύτερη, καλύτερη αντιμετώπιση των απατών. Οι τροπολογίες προβλέπουν επίσης ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μειώσει ή να αναστείλει <clears throat> τι προσωρινές ε, καταβολές χρημάτων ή προκαταβολέ προ τα κάτω μέλη και όταν θεωρεί ότι τα εθνικά ελεγκτικά συστήματα δεν είναι ενισχύ ή δεν είναι αποτελεσματικά ή αν παρουσιαστούν σοβαρές παρατυπίες και ε, δεν υπάρξει ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Δηλαδή, περιμένουμε από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις κατάλληλες ενέργειες. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ψηφοφορία. Νομίζω ότι έχετε όλη την κάρτα σας. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε όμως με ανάταση χειρών. Παράγραφος 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. δεικτή. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 εκπίπτει. Πάμε στην τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 Λάιον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δέκα υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δώδεκα υπέρ κατά αποχές δεκτή Τελική ψηφοφορία λοιπόν της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εντάξει. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το περιβάλλον μέχρι το 2020. Ευζοία στα όρια του πλανήτη μας. Η συγγήτρια κυρία Ντατσάνα Οκτάβια Σάρμπου. Δυστυχώς η κυρία Σάρμπου δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Θα την αντικαταστήσει ο ο Λουί Κάπουλο Σάντο, που είναι ο συντονιστή των Σοσιαλιστών. Αν δεν έχει να πει κάτι, Λουί, μπορούμε να προχωρήσουμε. Λουί. Μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσω, ε, κύριε Πρόεδρε. Απλώ έχω μια προφορική τροπολογία που ήθελα να παρουσιάσω, αλλά θα το κάνω στην κατάλληλη στιγμή. Καλά. Ευχαριστούμε, Λουί. Ξεκινάμε. Έχετε όλοι ε, τον κατάλογο ψηφοφοριών και την κάρτα σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με ανάταση χειρό. Αιτιολογική σκέψη 9, τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 1 του εισηγητή υπέρ κατά απόχες δεκτή 20 υπέρ κατά απόχες ε, πάμε στην 24 υπέρ κατά απόχες δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για 19, θέλετε, ναι, όχι, εντάξει. Έλεγχος για την 19. Άρχεται η ψηφοφορία. θα πρέπει να το κάνουμε με καταμέτρηση των ε, χειρών. Υπέρ της 19, σηκώστε τα χέρια σας. A Κατά. Εγκρίνεται. 19-17. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 19 σε ό,τι αφορά την παράγραφο 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 όχι. Όχι, όχι. Εκπίπτει. 22 υπέρ 22 Νταντέν υπέρ κατά από χέρι εγκρίνεται η 19 για την τέταρτη παράγραφο τέταρτη πρόταση είναι υπέρ κατά Εγκρίνεται. 20, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, εκπίπτει 20. 23. 23, υπέρ. Συγγνώμη, πρώτα η 24 πρώτα. 24. Σιλβέστρης, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο του εισηγητή υπέρ της εισηγήτριας μάλλον κατά Απόχες. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 25. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 26. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος. 28 υπέρ. <coughs> Okay. Okay. Adesso chi è contro le... Ποιος είναι κατά τις 28. Ε, Απορρίπτεται. Δεκα, 18, 18, 10 υπέρ, 18 κατά. 29 υπέρ. εντάξει, κατά. Απορρίπτεται με 12 εναντίον 18. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά Από Χέσεγκριντ. 32 υπέρ υπέρ κατά Απορρίπτεται. 10-16. 33. Γκάμπριελ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Είστε υπέρ, εντάξει. Κατά τώρα. Καλύτερα να μετρήσουμε. Δεκαέξι έντεκα γίνεται δεκτή, 34. Ο Μάρκ. Εγώ χαίρομαι για τη μεγάλη εσωτερική πειθαρχία τη ομάδα του ΕΛΚ, η οποία είναι αξιοσημείωτη. Αλλά αφού δεν έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, πρέπει να σηκώνουν όλοι τα χέρια του. Εγώ είδα να απορρίπτονται τροπολογίες όπου οι σοσιαλιστέ, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι ήταν μαζί. Λοιπόν, όλοι πρέπει να σηκώνουν τα χέρια του ώστε να δω πιο ψηλά για να γίνεται κατάλληλη καταμέτρηση. Δεν λέω για το παρελθόν, λέω για το μέλλον. Να σηκώνετε καλά τα χέρια σας για να φαίνεται, θα είναι σαφέστερο για όλους. Εντάξει, Μάρκ. Μα δεν δουλεύει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τι να κάνουμε. Μαρία, ε, δεν μπορούμε να βλέπουμε με αυτή την κάμερα τι γίνεται. Οκ. Emendamento, per favore, Silvestri. Εντάξει, 36. 35, συγγνώμη. Υπέρ. 35, υπέρ. Σηκώστε τα τα χέρια. 35. 35 Ποιοι είναι κατά παρακαλώ. Ε, τώρα το ΕΛΚ είναι πιο δυναμικό. Και οι φιλελεύθεροι βλέπω, ναι, ναι. Απορρίπτεται. 12-20. Πάμε στην 36. Υπέρ της 36. Κατά. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κα... Υπέρ, υπέρ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. 38. Κλάς Ρέιμες. Ε, εντάξει. Κατά. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. κατά εγκρίνεται. Πέντε. Πέντε συζητήτριες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα πέντε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα έξι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 της εισηγήτριας. Και εδώ ο Λουίς θέλει να πει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Να σας παρουσιάσω την προφορική τροπολογία, η οποία λέει τα εξής. Να μειωθούν μέσα σε, κατά πέντε χρόνια το χρονικό διάστημα που πρέπει να οδηγήσει σε μείωση 50% της σπατάλης τροφίμων και αυτό θα βοηθήσει να έχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα η απόφαση που έχουμε λάβει στην έκθεση Καρόνα για το ίδιο αυτό θέμα. Και όπου προβλεπόταν η ημερομηνία του 2025 και όχι 2030. Για λόγους συνεκτικότητας λοιπόν προτείνω να έχουμε την ίδια αυτή ημερομηνία και στο έγγραφο αυτό. Υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται στην προφορική τροπολογία. Ωραία. Οκτώ με αυτή την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 59 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 60 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 61 υπέρ. Να μετρήσουμε. Υπέρ. 61. Έχουμε τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάνουμε, αρχίζουμε την ψηφοφορία. 61 Πόλσεν και λοιπή. Άρχεται. Εντάξει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 64 υπέρ κατά απόχες δεκτή 65 υπέρ υπέρ κατά απόχες απέριπτε απορρίπτεται 9 τι Ήτρες υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 67 66 το τελευταίο τμήμα 66 φεϊμών τελευταίο τμήμα υπέρ 66 κατά αποχές απορρίπτεται 67 Αντρίου υπέρ κατά αποχές εγκριντ 68 υπέρ κατά αποχές εγκριντ 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κα, υπέρ υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τσεκ 72 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία ψήφισατε όλοι πέρας Απορρίπτεται 14-22. 10 υπέρ της 10. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές από... ναι. 75. Υπέρ. Κα... Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Κάνουμε έλεγχο για την 75. Για την 75. Άρχεται. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Για την 75. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται 14-20. 76 Λουκούμια ψηφοφορία. 76 Αντρίου. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Για τη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ και 4 αποχές καμιά ψήφο κατά. Συγχαρητήρια στην κητήρια Σάρμπα παρά την απουσία της. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 6. είναι ευρωπαϊκή ενίσχυση στους ε, πιο δύναμους. Ψηφίζουμε την έκθεση του συνεδέφου Μάρκ Νταραπέλε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση. Α, γαλλικά φαίνεται ότι είναι εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει το ρόλο. Δοκιμάστε. Εντάξει είναι τώρα, λειτουργεί. Καλώς. Ψηφίζουμε την έκθεση Μακταραμπέλα που είναι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πιο δυναμούς. Η αρμόδια Επιτροπή επί της ουσίας είναι η απασχόληση. Οι διάφορες ε, τροπολογίες. Υπάρχουν Τροπολογίε που έχουν καταθέσει οι βολευτές και προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική ψηφοφορία υπάρχουν συμβαστικέ τροπολογίε που ετοίμασαν οι συνάδελφοι, ο Ταραμπέλα και οι σκιώδες εισηγητέ μαζί. Μάρκ, θέλεις να εξηγήσει λιγάκι. Ναι. Πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ τη γραμματεία, η οποία ανέβαλε για μία εβδομάδα την ψηφοφορία. Και έτσι μπορέσαμε να έχουμε κάποιους συμβιβασμούς. Συμβαστικές τροπολογίες που θα έλεγα ότι δεν αποτελούν αντικείμενο μιας απόλυτης συμφωνίας, αλλά μη τι άλλο διάφορες επιμέρους τροπολογίες έτσι έχουν βγει από το τραπέζι. Πρόκειται είτε για ποσά, ο λόγο είναι ότι δεν θέλουμε να βαρύνει πολύ το ταμείο αυτό και να μπορέσει έτσι να επιβιώσει και να εξυπηρετήσει μια Ευρώπη μέσα στην οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη από επιστημιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τις πολιτικές ομάδες για την εξαιρετική τους βοήθεια. Όσες τροπολογίες βέβαια δεν μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες, ελπίζω να είναι λίγο πολύ κατανοητές και να μπορέσετε να τις εγκρίνετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μάρκα. Συναδελφοί, έχουμε πολύ μεγάλη ψηφοφορία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Διανατάσεις χειρός. Ας ε, προχωρήσουμε και μετά θα δούμε τι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Όχι, 7 διορθώνει ο πρόεδρο. 7. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. 11-16. Θα ελέγξουμε όμω για να είμαστε σίγουροι. Πρόκειται για την τροπολογία 7. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 16 κατά. Διανατάσσεως στις χειρός τώρα. 77. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Όχι. Όχι, αποσύρεται αυτή. 70. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. <clears throat> Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Όχι, έχει εγκριθεί αυτή. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. 83 υπέρ. 83 κατά τώρα. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Όλοι κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 τώρα μπέλα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 λεμπρά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 Ολέτσνικα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93, Αντρέα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94, υπέρ, 94, υπέρ, κατά, Θα ελέγξουμε για την 94 του κύριου Αντρία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 19-16. Τώρα, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία αριθμός 2. Α, όχι, αντιανατάσσεως της χειρός. Ποιοι είναι υπέρ της συμβαστικής 2, παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 Μποβέ υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε για την 95 του κυρίου Μποβέ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 16-17. Τροπολογία 97 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 Αντρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκατόν εννέα, Νικουλέσκου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Να σηκώνετε καλά το χέρι για την 113 μαγκίνες. Υπέρ. Υπέρ 113. Κατά. Εγκρίνεται. 115. Λεμπρά. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Και δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε για την 115 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 18 υπέρ 17 κατά. 116 υπέρ. Κατά. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε για την 116. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τις ψηφοφορίες. 16 υπέρ, 19 κατά απορρίπτεται. 117 υπέρ, διανατάσσεως χειρός, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 121. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Όταν είναι τόσο σφιχτό το αποτέλεσμα πρέπει να ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά λοιπόν ελέγχουμε για την 122. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 18-17 το αποτέλεσμα εγκρίνεται. 123. Υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Είχα να προτείνω κάτι, Πρόεδρε. Όταν βλέπετε ότι το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές, που είναι οι πιο μεγάλες ομάδες, διαφωνούν, τότε αμέσως να λέτε ηλεκτρονική ψηφοφορία για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος, θα ακολουθήσουμε τον εισηγητή. Συνεπώς, ο Ταραμπέλα που είναι εισηγητής και ο σκιώδης του ΕΛΚ να μου δείχνετε. Όταν βλέπω ότι διαφωνείτε μεταξύ σας θα λέω αμέσως ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εντάξει. Ποιο είναι, σε Α, εκείνη. Α, ωραία, για να ξέρω πού να κοιτάω. Α, εντάξει. Ωραία. Καλώ. 123 ε, αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18-16. 124 υπέρ. Να δω. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 124. Ψηφίσατε όλοι. Για την 124 πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. 125. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 126 τώρα. Υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για την 126. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 127 υπέρ. Υπέρ 127 κατά. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την 127. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας προφορίες. Ισοψηφία. Που σημαίνει ότι απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 129. Τι, όχι. 130 τώρα. 130. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ για την 130. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 132 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ για την 133. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 134 Νικουλέσκου υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 134. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Σικυρέσκι, τι ψηφίζετε, όλοι σα κοιτάνε. 135. Κατά. Ωραία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Για την 135 ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 136. Υπέρ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την 136. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. 136. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. 138. Κατά. Α, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 138. Ψηφίστε παρακαλώ. Λοιπόν, μια στιγμή. Θα ψηφίσουμε μαζί 138 με 144. Αν μπλοκ όλες μαζί δηλαδή αυτές οι τροπολογίες με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 138 μέχρι και 144. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνονται. 138 με 144. Τώρα, 145 υπέρ, ηλεκτρονικά. Καλώς. Τις τρεις τροπολογίες Νικουλέσκου μαζί τις ψηφίζουμε. 145. Δεν γίνεται. 145 τότε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία για την 145. Εγκρίνεται. 146. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 146. Πέρα τη εγκρίνεται. 147 τώρα. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 148. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 148. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 149. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 149. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 151. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίνεται. 152. Υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 152. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 153. Μάρκ, τι είσαι κατά. Α, ηλεκτρονικά λοιπόν για την 153. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 155. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 155 εγκρίνεται. Τώρα. 156. Υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 156. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 156 απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 158 Νικουλέσκου. Κατά. Βλέπω. Κατά. Ποιο είναι κατά. Απορρίπτεται. 159. Υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 159. Πέρες προφορίες. Εγκρίνεται. 161. Υπέρ. ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την 161. Ψηφίστε. στις της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 162 Νικουλέσκου. Η... Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 162. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίνεται. 163. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 163. Ψηφίστε. Α, Μάρκ. 163 ε, εγκρίνεται, αλλά το λόγο έχει τώρα ο Μαρκ Ταραμπέλα. Οι τροπολογίε αυτέ ψηφίζονται δημοκρατικά, είναι μια απλοποίηση βασικά του κειμένου τη Επιτροπή. Και ναι, μεν συμφωνώ με όλε τι τροπολογίε που προτάθηκαν από του κύριους Λαμπρά κλπ. Παρ' όλα αυτά, διαφωνώ και λέω στην ομάδα μου να καταψηφίσει για εκείνες όπου οι διατάξεις ε, έτσι εξαφανίζονται. Όλοι θέλουμε απλοποίηση. Το ζήτημα είναι ότι εξαφανίζονται κάποια πράγματα. Βέβαια, επειδή δημοκρατικά ψηφίζουμε, ζητάω από την ομάδα μου να ψηφίσει. Θα είναι μια απλοποίηση του κειμένου, θα είναι θετικό, ο κίνδυνος βέβαια είναι, γι' αυτό και εγώ έβαλα μείον σε διάφορες από αυτές τις τροπολογίες, γιατί ναι, μεν ε, θέλουμε απλοποίηση, αλλά δεν θέλουμε να εξαφανίσουμε. Λοιπόν, προτείνω να υπερψηφίσουμε όμως τώρα, είναι έτσι κι αλλιώς ξεκάθαρο ποια είναι η πλειοψηφία εδώ, οπότε για να απλοποιηθεί η ψηφοφορία το λέω δηλαδή. Δηλαδή, ωραία, αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Εντάξει, ωραία. Είμαστε στην 164. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 Ολενίτσεκ. Υπέρ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για το 176. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. ο χειρό. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 182. Λεμπρά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ο εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 186. Νικουλέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187. Υπέρ. Υπέρ. Α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 187. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 188 λεμπρά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 αντάτη υπέρ. Α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 189. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. 190 Νικολέσκου υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 190. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 14 του συγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μια στιγμή. No, 193. 193. 193. Σάρβου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 Νταντσίλα υπέρ, κατά, α, όχι, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για την 196. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες για την 196. Εγκρίθηκε. 15 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. «201. Πατρών υπέρ». Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το 201. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 202 λεμπρά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 Νικουλέσκου υπέρ. Α, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 206. Ψηφίστε παρακαλώ. 205, 205. Όλοι ψηφίσατε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τώρα 206 λεμπρά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε μαζί από τη 207 μέχρι τη 222. Συμφωνεί ο συγγετής, οι ομάδες, συμφωνείτε, ωραία. Ψηφίσουμε μαζί όλες αυτές τις τροπολογίες ηλεκτρονικά. Α, όχι. περ κατά, αποχές, εντάξει, αφού συμφωνείτε όλοι, εγκρίνονται έτσι. Και φτάνουμε Μια που είναι όλοι οι ομάδε, γι' αυτό αποφάσισα τελικά να ψηφίσουμε ω χειρό, λέει ο πρόεδρο. 224. 224 υπέρ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. 224. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα, Συμφωνούμε όλοι να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες από 222 λεμπρά, α, 225 γιατί την ψηφίσαμε τις προηγούμενες, 225 λοιπόν από την 225 μέχρι τη 262 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίθηκαν. Ωραία. 263 τώρα τα ραμπέλα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 265 λεμπρά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200... Α, όχι. Αιτιολογική σκέψη 17 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, α, ηλεκτρονικά. Αιτιολογική σκέψη 19. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 20 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 21. Ψηφίσατε όλοι. περασε της προφορίας. Απορρίφθηκε. 22 υπέρ. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 22. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 23. Γκουλάρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Λεμπρά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Μποβέ. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 26. Υπέρ. Κουλάρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 του υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 34. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. 35 λεμπρά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 Ντάνσιλα υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 36. Ψηφίστε παρακαλώ. Όλοι είναι κατά, ε. Α, πέρα στις ψηφοφορίες απορρίφθηκε. Μαρκ, να μην ε, χασομεράμε. 37 λεμπρά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 λεμπρά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 κουλάρι υπέρ. Α, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 43. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 17-17. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 5. Του εισηγείται υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45. Μποβέ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Λεμπρά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 γκουλάρι πέρ. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για τη 47. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Πάλι με ισοψηφία. 17-17. 48 λεμπρά υπέρ. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 λεμπρά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 λεμπρά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 τώρα λοιπόν Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 τάντσιλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέλος 62 υπέρ Λεμπρά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροποποιημένη γνωμοδότηση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα της οφορίας, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε Μάρκ Ταραμπέλα συγχαρητήρια. 27 υπέρ 3 κατά και 4 ε, αποχές. Ε, συγχαρητήρια κύριε Ταρά Μπέλα. Ο κύριος Ταμπάζδη που είναι. portare l'ultimo che disse noi due minuti che ha fatto. Ευχαριστώ. Dai colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε στο τελευταίο θέμα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή. Το 6 λοιπόν, επεξεργασία, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού με εισηγητή γνωμοδοτήσεως τον κύριο Ταμπάζντι. Ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση οδηγίας της Κομισιόν για την εναρμόνιση των διαφόρων διατάξεων στις χώρες μέλη σχετικά με την επεξεργασία, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων. Ο συνάδελφός μας κ. Σταμπάζντι θα συντάξει γνωμοδότηση για λογαριασμό μας και παρακάλεσε να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν. Από την Γενική λοιπόν Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχουμε την εκπρόσωπο κυρία Βήμαρ η οποία θα προβεί σε ανάπτυξη της προτάσεως της Κομισιόν και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Νταμπάζη. Θα παρακαλέσω λοιπόν την εκπρόσωπο της Κομισιόν να λάβει πρώτη αυτή το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για την, για την ε, ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να αναπτύξουμε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία περί προϊόντων καπνού. Το Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη έχει ζητήσει να υποβληθεί πρόταση από την Κομισιόν για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για προϊόντα καπνού εποφελία των Ευρωπαίων πολιτών. Τον Δεκέμβριο του 2012 εγκρίθηκε τελικά από την Κομισιόν η πρόταση μετά από μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων και στην βάση σε βάθος μελέτης επιπτώσεων. Ο λόγος για την αναθεώρηση της τρέχουσας οδηγίας ήταν προφανής. Η νομοθεσία αυτή είναι ήδη 12 ετών και δεν συμβαδίζει πλέον με τη σημερινή πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αγορά, επίσης τις επιστημονικές και διεθνείς εξελίξεις. έχουν εμφανιστεί νέα προϊόντα καπνού στην αγορά, τα οποία μοιάζουν σαν ε, κραγιόν των χιλιών, έχουν διάφορες γεύσεις, ε, βανίλιας ή άλλα και ε, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά ιδίως για τους νέους. Επίσης οι χώρες μέλη έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τα ίδια αυτά, κάτι το οποίο οδηγεί σε κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς. Επίσης, υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα, για παράδειγμα για τις προειδοποιήσεις υγείας. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες μέλη της έχουν συνυπογράψει την, τη συνθήκη πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο των πρώτων καπνού που, ε, που εφαρμόζεται από το 2005 και εμείς έχουμε πλέον εκ του νόμου υποχρέωση να ε, συμμορφωθούμε με τις διατάξεις της. Η πρόταση της Κομισιόν στοχεύει ιδιαίτερα στους νέους και σε μέτρα αποτροπής τους από το να αρχίσουν το κάπνισμα ή την κατανάλωση καπνού. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι 70% των καπνιστών αρχίζουν σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Και σχεδόν κανείς δεν αρχίζει το κάπνισμα μετά τα 25 χρόνια της ηλικία. Άρα μιλούμε για πραγματικά νέους. Οι νέοι αρχίζουν το κάπνισμα διότι το βρίσκουν cool και αργότερα συνεχίζουν διότι βεβαίως έχουν εφιστεί. Με τα χρόνια το κάπνισμα οδηγεί σε καρδιακές παθήσεις, καρκίνους και ένα σωρό άλλα προβλήματα υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα για 700.000 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο λόγω εξαιτίας του καπνίσματος. Εντελώς περιττή θάνατη. Εκτός όμως από τη θνησιμότητα, ο καπνός, το κάπνισμα προκαλεί χρόνια δεινών, παθήσεων και βεβαίως τεράστια δημόσια δαπάνη. Πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και αυτά είναι και μετριοπαθείς υπολογισμοί. Επίσης υπάρχουν και άλλοι έμεση κίνδυνοι όπως απώλεια της αναπαραγωγικότητας. Επίσης ζημία για την κοινωνία. Για αυτούς τους λόγους θεώρησε η Κομισιόν ότι πρέπει να επιβληθούν κάποιες ρυθμίσεις στα προϊόντα καπνού ώστε ο κόσμος να ξέρει τι αγοράζει και ότι αυτό που αγοράζει είναι ένα επικίνδυνο εθιστικό προϊόν. Τι προτείνει τώρα η Κομισιόν. Θα ήθελα να αρχίσω από την επισήμανση έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν με κάποια ενημέρωση. Η πρόταση προβλέπει μεγάλες υποχρεωτικές εικόνες που θα καλύπτουν 75% του μπροστινού και το πίσω μέρος του πακέτου των τσιγάρων. Και στα πλάγια πάλι επίσης επισημάνσεις υγείας. Επίσης η πρόταση δεν επιτρέπει διαφημιστικά στοιχεία ε, προϊόντων καπνού που να είναι ελκυστικά για τους νέους. Για παράδειγμα, πακέτα όπως αυτό που να μοιάζει σαν lipstick, σαν κραγιόν ε, χιλιών, σαν αυτό που σας δείχνω εδώ, δεν θα επιτρέπονται πλέον. In Τις τελευταίες εβδομάδες δεχθήκαμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πόσο ποσοστό του πακέτου θα είναι ρυθμισμένο και πόσο θα είναι ελεύθερο, ελεύθερη χρήση. Εμείς ε, προβήκαμε στους μαθηματικούς υπολογισμούς και εάν συμπεριλάβετε όλες τις επιφάνειες, περίπου 30% του πακέτου εξακολουθεί να είναι ελεύθερο για τις χώρες μέλη ή για τα εμπορικά σήματα αναλόγως. Από την άλλη μεριά η πρόταση επιτρέπει στις χώρες μέλη ε, να προχωρήσουν περισσότερο και να ε, εφαρμόσουν, να επιβάλλουν δηλαδή τα απολύτως σκέτα πακέτα τσιγάρων, το plain packaging. Τώρα, ένα μέρος της προτάσεως αναφέρεται στα συστατικά του καπνού. Προβλέπει τα πρόεδρα του καπνού με ειδικέ γεύσεις, όπως ας πούμε βανίλια ή μεντόλ, να μην επιτρέπονται. Διότι αυτά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους και τις νέες και διευκολύνουν το να αρχίσει κανείς να καπνίζει. Επίσης, ενδεχόμενα παραπλανητικά, παραπλανητικές ενδείξεις όπως για παράδειγμα καφεΐνη ή βιταμίνες. Επίσης δεν θα επιτρέπονται στα προϊόντα καπνού. Η πρόταση, και θα ήθελα εδώ να το τονίσω αυτό, η πρόταση δεν ρυθμίζει τα πρόσθετα τα οποία είναι ίσως απαραίτητα για την παραγωγή προϊόντων καπνού, όπως για παράδειγμα η ζάχαρη, που είναι απαραίτητη που προστίθεται σε ορισμένα καπνά για να αποκαταστήσει την ποιότητά τους. Που ένα ποσοστό της ζάχαρης χάνεται από την ξύρανση των φύλων καπνού. Δεν κάνει και διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών καπνού, ούτε αποτρέπει την διαφοροποίηση των διαφόρων ε, μαρκών εφόσον δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ισχυρή διαφοροποιητική γεύση. Α έρθω τώρα σε, άλλες άλλα θέματα τη προτάσεω. Όσον αφορά τον καπνό σνούζ, η πρόταση προτείνει τη διατήρηση του status quo, δηλαδή να παραμείνει η απαγόρευση του σνούζ στην Ευρώπη, εκτός από τη Σουηδία, η οποία διατηρεί εξαίρεση. Με την επιχειρηματολογία ότι το σνούζ είναι εθιστικό, έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία και δεν υπάρχει δεν υπάρχουν πραγματικέ ενδείξεις ότι όντω βοηθάει τον κόσμο να, να αφήσει το κάπνισμα, να σταματήσει το κάπνισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που είναι πάλι καινούργια εξέλιξη, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι προϊόντα με ένα περιεχόμενο νοικοτήνη πάνω από κάποιο κατόφλι θα πρέπει να ε, είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν έγκριση όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό είναι ήδη η ε, κατάσταση που ισχύει σε πάνω από τις μισές χώρες. Αυτά που έχουν λιγότερη νοικοτήνη κάτω από το κατόφλιο δηλαδή, μπορούν να πολλούνται ελεύθερα στους καταναλωτές εφόσον φέρουν τις απαραίτητες επισημάνσεις. Θα πρέπει να γράφουν επίσης απάνω nicotine replacement therapy και διάφορα τέτοια και να ανταποκρίνονται σε ένα πλαίσιο μέτρων προφύλαξης ειδικά για τα προϊόντα αυτά. Τέλος, μια παρατήρηση για το παράνομο εμπόριο. Η Κομισιόν στην πρότασή της προβλέπει λήψη ισχυρών μέτρων κατά του παράνομου εμπορίου και ένα σύστημα δηλαδή χνηλασιμότητας και ανείχνευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα καπνού, καθώς και ορισμένων ενδείξεων ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού. Μέτρα τα οποία θα προστατεύουν τους πολίτες απέναντι στα παράνομα προϊόντα και ταυτόχρονα θα προστατεύουν και τους νόμιμους προμηθευτές και εμπόρους καπνού πολλοί από τους stakeholder στις διαβουλεύσεις μας εξέφρασαν ανησυχίες για το παράνομο εμπόριο και γι' αυτό προτείνει η Κομισιόν αυτά τα αποτελεσματικά μέτρα τα οποία συμμορφώνονται απολύτως με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις και τις εξελίξεις στον χώρο. Τέλος, μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, για τις επιπτώσεις της, προτάσης, της προτάσεως. Καμιά φορά ακούγονται γνώμες που λένε ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις η πρόταση στους παραγωγούς καπνού ή στη βιομηχανία καπνού. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι καθόλου δραματική η προβλεπόμενη επίπτωση της οδηγίας. Προβλέπεται για πέντε χρόνια 2% μείωση του αριθμού των καπνιστών. Αυτό προβλέπει η Κομισιόν. Αυτό σημαίνει 2,4 εκατομμύρια καπνιστές λιγότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σωθούν πολλές ζωές, δεν θα συνεπάγεται όμως δραματικές αλλαγές για τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπόριο του καπνού. Επίσης, το κόστος για την καπνοβιομηχανία θα μετριαστεί από τα μέτρα που θα ληφθούν κατά του παράνομου εμπορίου και θα εξισορροπηθεί και από τις ωφέλειες που θα προκύψουν από την αυξημένη εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Στην απασχόληση οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι συνολικά θετικές, διότι τα χρήματα τα οποία δεν θα δαπανά ο καταναλωτής για την αγορά προϊόντων καπνού, θα τα δαπανά η αγορά άλλων προϊόντων και άλλων υπηρεσιών, που είναι λιγότερο εντατικές εργασίες. Και εν τέλει, όπως είπε και ο Πίτροπος Μπόρς, η πρόταση της Κομισιόν είναι φιλόδοξη αλλά ισορροπημένη και η Κομισιόν επιθυμεί να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο για να προχωρήσει σύντομα στην υιοθέτηση αυτής της σημαντικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την δόκτωρα Βίλμερ. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον Τσάμπα. Τι προτιμάτε Τσάμπα εσείς, ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο θέμα και η πρόταση φυσικά είναι πολύπλοκη και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή κύριε Πρόεδρε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και γνωρίζω πολύ καλά τις διαμάχες που αφορούν το θέμα αυτό. Μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκρουση μεταξύ της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Γεωργίας για το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι σαφές στο μυαλό μας είναι ότι έχουμε ένα κοινό στόχο να εξασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Θέλουμε να υπάρξει μία μείωση του αριθμού των καπνιστών μεταξύ των νέων Και εδώ θα πρέπει να πω προς τα μέλη της Επιτροπής μας ότι τα επιχειρήματα τα οποία εγώ ανέπτυξα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα τα αναφέρω και εδώ μιλάμε για 400.000 γεωργούς και φυσικά μετά από τη δημόσια υγεία η δεύτερη μας προτεραιότητα είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να, για να διατηρήσουμε τους ε, καλλιεργητές αυτούς που ζουν στις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 96% από αυτούς είναι μικρογεωργοί, που έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις μεταξύ μισού και τριών εκταρίων. με την εισηγεσία του κυρίου Παπαστάμκου, η δική μας Επιτροπή έχει τονίσει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της παραγωγής καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της επεξεργασίας, της μεταποίησης του καπνού. Η μεταποίηση καπνού στην Ευρώπη χρησιμοποιεί μόνο 25% κατά 25% του καπνού ο οποίος ε, παράγεται στην Ευρώπη. Δηλαδή το 1 πέμπτο μονάχα του καπνού που μεταπείται στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Επομένως, στην ε, έκθεση αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε και την απόλυτη ανάγκη να διατηρήσουμε τη θέση εργασίας στη Γεωργία και υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει το, η διάπτωση των τιμών με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεγάλες μεταποιητικές εταιρείες θα αποσυρθούν από την Ευρώπη και θα παίρνουν καπνό από φτηνότερους παραγωγού καπνού, παραγωγούς καπνού σε τρίτες χώρες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή μας συγγνώμη, από την Εθνική Επιτροπή συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας να προβεί σε μια έκθεση αντικτύπου. Να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος ο οποίος θα προκύψει για τις τιμές και την κερδοφορία και τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα επηρεάσουν την κατάσταση των 400.000 καπνοπαραγωγών. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ε, υπεύθυνο από τη δική μας πλευρά να πάρουμε μια απόφαση χωρίς έκθεση αντικτύπου και για, τον, για το κάπνισμα στους νέους. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς οι οποίοι θέλουν να μειωθεί η χρήση καπνικών προϊόντων μεταξύ των νέων. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια προληπτική πτυχή την οποία θα ενισχύσουμε μέσω, αυτή την, μέσω αυτής της πρότασης. Εγώ θα ήθελα να δημιουργήσουμε ένα ταμείο για την πρόληψη του καπνίσματος Κάτι τέτοιο υπάρχει στη Γερμανία και το γερμανικό παράδειγμα είναι παράδειγμα προς Γιατί δείχνει ότι σε μια χώρα όπου γίνονται σοβαρές προσπάθειες πρόληψης υπάρχει πράγματι μείωση του αριθμού των καπνιστών. Αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται και στη Γαλλία, όπου γίνονται προσπάθειες να μειωθεί η πρόσβαση σε καπνικά προϊόντα. Στην ε, Γαλλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία υπάρχει ένα όριο ηλικίας 16-18 ετών κάτω από το οποίο δεν μπορεί να αγοράζει κανείς καπνικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και επίσης για τις πωλήσει μέσω διαδικτύου εγώ εντυπωσιάζομαι που βλέπω δεν υπάρχει καμιά απαγόρευση για την πώληση καπνικών προϊόντων στο διαδίκτυο, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να πολλούνται τα καπνικά προϊόντα στο διαδίκτυο, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η πρόσβαση που έχουν οι νέοι στα προϊόντα αυτά και αυτός είναι εξάλλου ο κύριος στόχος μας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι οι καπνιστές ξεκινάνε το κάπνισμα πριν από τα 25. 98 περίπου τα 100 όλων αυτών που καπνίζουν ξεκινήσαν το κάπνισμα πριν από τα 25. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε στους νέους. Και υπάρχει και μια άλλη σημαντική πτυχή. Στην προηγούμενη οδηγία για τα καπνικά θέματα, ο καπνός θεωρήθηκε ότι είναι μονάχα ένα συστατικό, ένα, μάλλον ένα συντελεστής και όχι ένας όχι ένα συστατικό. Υπάρχει αυτή η ίδια ε, διαμάχη για τους συντελεστές και τους, τα συστατικά στην οδηγία για τη γύρη και το μέλλον. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να έχουμε μια διατύπωση που δεν θα μας εκθέσει σε νομικές διαμάχες. Εγώ έχω νιώσει ότι μας έχει υποστηρίξει η Κομισιόν <clears throat> ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, παραγωγή καπνού Burley, από καπνά Burley, προσθέτοντας ζάχαρη κατά τη διαδικασία της ξύρανσης και επεξεργασίας του καπνού. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αυτή η εγγύηση για τους παραγωγούς του καπνού από καπνά Burley. Για τις προσθετικές ουσίες, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να απαγορευτούν αυτές οι ουσίες που δίνουν ειδικά ειδικέ γεύσει όπω η βανίλια, η σοκολάτα, η καφέινη, όλα αυτά πρέπει να απαγορευτούν. Η καφέινη και οι βιταμίνες πρέπει να απαγορευτούν γιατί έχουν ένα παραπλανητικό χαρακτήρα. Αν έχετε ένα προϊόν που έχει την επιγραφή ότι περιέχει βιταμίνες, αυτό είναι παραπλανητικό και δεν πρέπει επομένω να επιτραπεί. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε ένα θετικό κατάλογο και σε ένα αρνητικό κατάλογο. Εγώ δεν βλέπω στην τωρινή πρόταση να υπάρχουν <clears throat> τέτοιοι κατάλογοι. Και η μέντα είναι ένα ειδικό θέμα το οποίο αναφέρθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για την μέντα, το μενθόλ, οι περισσότεροι υποστηρίζουν την απαγόρευσή του. Λένε οι πολλές ε, ιατρικές μελέτες ότι το δροσιστικό αποτέλεσμα του μενθόλ οδηγεί σε βαθύτερη εισπνοή καπνού. Υπάρχουν όμως ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία, όπου τα τσιγάρα με μέντα είναι παίζουν σημαντικότερο ρόλο, έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Και ίσως θα πρέπει να δούμε και το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, όπου στις χώρες αυτές, σε αφότερες τις χώρες αυτές, επιτρέπεται η χρήση μενθόλης για να παίρνουν γεύση τα τσιγάρα. Δεν λέω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο, απλώς θέτω αυτό το ερώτημα. Τώρα, για όλα αυτά τα οποία έχουν ε, που φαίνονται σαν κραγιόν, σαν γυναικείο κραγιόν, <clears throat> αυτό είναι πραγματικά απόλυτα παραπλανητικό. Και επίσης αυτά τα τσιγαρλίκια τα οποία μοιάζουν με σοκολάτα, τα πουράκια που είναι σαν σοκολατένια πουράκια, μπορούν να δημιουργήσουν και αυτά μια παραπλάνηση στους νέους. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Η συσκευασία σε κουτιά χωρίς καθόλου σήμανση και διαφημίσεις είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε. Εδώ βλέπετε ένα πακέτο το οποίο είναι σε μια συσκευασία απόλυτα σκέτη, απλώς υπάρχει το όνομα της εταιρεία στο τέλος και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι προειδοποίησεις για την υγεία υπάρχει υποστήριξη για μια τέτοια συσκευασία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και πιστεύω και εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, λύση αυτή. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας σε σχέση με τέτοια συσκευασία. Δεν έχουν αρκετές πληροφορίες σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση γιατί δεν αναφέρονται η, η περιεκτικότητα σε πίσα, ο μονοξίδιο του άνθρακος κτλ. Αυτό μπορεί να είναι πράγματι παραπλανητικό. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς ποια τσιγάρα είναι πιο βλαβερά. Όλα είναι βλαβερά βέβαια, αλλά οι καταναλωτές θα έχουν μεγάλη δυσκολία να τα συγκρίνουν από την πλευρά αυτή. Επομένω, εδώ τίθεται ένα θέμα προστασία καταναλωτών για τα εμπορικά σήματα επίσης. Υπάρχουν σήμερα θέματα στα οποία δεν πρέπει να επισέλθουμε σε Επιτροπή Γεωργίας. Εμείς θα πρέπει να σταθούμε μονάχα στα θέματα υγείας και στα θέματα των καπνοπαραγωγών τα θέματα των ηλεκτρονικών ε, σιγαρέτων και των σημάτων, των εμπορικών σημάτων, δεν θα πρέπει να μας απασχολήσουν επομένω. Τέλος, εν κατακλείδη. Ένα πρόβλημα ακόμα, το οποίο είναι ένα, ένα θέμα που ανα, ανατρέχει σε πολύ παλιότερες εποχή, εποχές, το θέμα των ε, κατεξουσιοδότης πράξεων και των εφαρμοστικών πράξεων. Η πρότασή μου έχει ως εξής. Ας δούμε τον αριθμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων, που είναι πάρα πολλές αυτές οι οποίες δίνουν αυτή τη δυνατότητα στην Κομισιόν να δράσει. Αν δώσουμε αυτή την εξουσιοδότηση στην Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα αρνησικηρίας πάντα, να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να αποφασιστούν στο μέλλον. Και τέλος, να σας πω προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ αναφερθεί. Υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ του επίπεδου παιδείας και της χρήσης καπνικών προϊόντων, του καπνίσματος. 45% των ανδρών που έχουν μονάχα απολυτήριο δημοτικού καπνίζουν κάθε μέρα, ενώ μόνο 25% των Ευρωπαίων καπνίζουν. Αλλά, σας είπα και πάλι, 45% των ανδρών αποφύτων δημοτικού καπνίζουν. Ενώ αυτό το ποσοστό πέφτει για αυτούς που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Για είναι και είναι διαφορετικό. 26% για απολυτήριο δημοτικού, ε, λυκείου και πανεπιστημιακό πτυχίο. 26% και καταλήγει στα 18%. Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος ότι με την νέα συσκευασία, οι πιο τροτές κοινωνικές ομάδες θα έχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα πληροφόρησης σε σχέση με τους κινδύνους του καπνού, τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Επομένως, εν κατακλείδη, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καπνοπαραγωγούς, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος του να δώσουμε την εντύπωση ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ε, των καπνοβιομηχανιών. Είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία, είναι σχεδόν ένα είδος σχηνοβασίας, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή μας, τον κύριο Τσάμπα Ταμπάτζη, για την ε, προετοιμασία. Έκανε πάρα πολύ δουλειά. Τα συμπεράσματά του, αναμφίβολα, είναι πολύ καλά. Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση τώρα. Έχουμε πολλούς που έχουν ζητήσει το λόγο και θα αρχίσουμε με τον κύριο Σκοτά και μετά τον κύριο Μποβέ. Παρακαλώ, Σκοτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, εγώ σας ε, επιβεβαιώνω ότι εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμών ε, στην Επιτροπή εδώ Γεωργίας πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με τέτοια προϊόντα όπως είναι τα καπνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Είμαι υπέρ μιας πολιτικής η οποία να ενισχύει ακόμα περισσότερο την καταπολέμηση της συνήθειας του καπνίσματος. Κάθε φορά που βλέπουμε μια βία εικόνα, όμως έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούμε. Το γεγονός ε, λοιπόν το ότι ζητάμε να μην καπνίζει ο κόσμος θα έπρεπε να φτάνει. Εγώ τώρα θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στην πρόταση αυτή οδηγίας και πιο συγκεκριμένα να μιλήσω για το ηλεκτρονικό αυτό σιγαρέτο. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία περιέχουν νικοτίνη. Το ηλεκτρονικό αυτό σιγαρέτο δεν μπορεί όμως να κυκλοφορήσει εμπορικά. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να διευρύνουμε τον έλεγχο ή το πεδίο εφαρμογή του άρθρου αυτού 18, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα προϊόντα που περιλαμβάνουν νοικοτίνη. Πολύ συχνά, βέβαια με ρωτάνε τι είναι τελικά. Είναι μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό τσιγάρο ή τελικά κάνει τους μη καπνίζοντες να θέλουν να καπνίσουν. Υπάρχουν ε, διάφορα είδη νικοτίνης, διάφορα είδη τέτοιου είδους σιγαρέτου, κάτι το οποίο προκαλεί μάλλον ε, σύγχυση στο μυαλό των καταναλωτών. Το ποσοστό περιεκτικότητας σε νοικοτήνη λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά αυτά σιγαρέτα που περιέχουν ε, νικοτίνη, να θεωρούνται θεραπευτικά. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια μελέτη περισσότερο σε βάθος για τους κινδύνους που ελοχεύει η χρήση τέτοιων ε, ηλεκτρικών ε, σιγαρέτων πριν αποφασίσουμε για την ε, εμπορία διαφόρων τύπων τέτοιων σιγαρέτων. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πώς δουλεύουν, τι κινδύνους ελοχεύουν, αλλά να κάνουμε και μελέτε σε βάθος, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τίποτα το τοξικό ε, από τη χρήση τους. Να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι ακριβώς οι επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Μπορεί να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Στην Βραζιλία απαγορεύονται αυτά τα τσιγάρα περιμένουν πρώτα να έχουν πιο συγκεκριμένα δεδομένα για το πόσο επικίνδυνα είναι. Ενώ στην Ιταλία τα ηλεκτρικά αυτά τσιγάρα πολλούνται άνετα, απαγορεύονται μόνο στους νέους κάτω των 16 ετών. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα έπρεπε να εξετάσουμε, το φορολογικό για παράδειγμα. Ίσως θα μπορούσαν κάποια μέρα να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά τσιγάρα Αυτοί όμως οι οποίοι θα διαφερθούν περισσότερο θα εμβαθύνουν περισσότερο και στο φορολογικό. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα της ε, βιομηχανίας καπνού. Και εδώ θα έπρεπε να αλλάξουν οι διατάξεις και να λάβουμε υπόψη μας την χρήση αυτών των νέων προϊόντων αν σήμερα χρησιμοποιούσαν πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο για παράδειγμα, τι θα κάναμε, δεν θα το απαγορεύαμε, γιατί δεν είναι πραγματικό τσιγάρο, είναι ένα gadget. Που όμως έχει διάφορες χημικές ουσίες. Ποιος θα με εμπόδιζε να το καπνίσω αυτό το ηλεκτρικό σιγαρέτο. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να γίνει μελέτη για την χρήση αυτών των ε, ηλεκτρικών τσιγάρων πέρα από την νοικοτήνη που περιλαμβάνουν. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως οι πιο νέοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Πρόεδρο, ευχαριστώ να τηρείτε το χρόνο σα, γιατί όπω ξέρετε έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση των συντονιστών με του Σκιώδη για τέσσερι εκθέσει που έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΠ ο αντιπρόεδρος Μποβέ, μετά Κορέα και Κλάς. Ο κύριος Μποβέ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω από τη δικιά μου την πλευρά ότι η συζήτηση αυτή ξεπερνάει πολύ το ρυθμιστικό πλαίσιο. Όλοι θυμόμαστε την αρχή, πώς αρχίσαμε να εξετάσουμε την οδηγία αυτή το 2009 και ότι ένα από τα σημαντικά συμβάντα της περίοδου αυτής ήταν ότι καθαρέθηκε ο αρμόδιος επίτροπος για το θέμα αυτό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν είναι ανεξάρτητο αυτό από την προσπάθεια που κάνουν πολλές μεγάλες εταιρείες να καθυστερήσουν την οδηγία αυτή. Να μην καταλήξει δηλαδή πριν τη λήξη της κοινοβουλευτικής μας Συνεπώς, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαψεύσουμε ακριβώς τις εταιρείε αυτές το κείμενο να εγκριθεί πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαι πεπισμένο ότι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ε, του καπνού κάνουν ό,τι μπορούν και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την έγκριση της οδηγίας αυτής. Οπότε πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πριν λήξει η θητεία μας. Και δεν είναι εύκολο. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις αυτές ε, φτιάχνουν και βρίσκουν καινούρια προϊόντα, εφεύρουν νέα προϊόντα, τα οποία τα συγκαταλέγουν σε μία κατηγορία και έτσι προσπαθούν να πολλούν προϊόντα παράγωγα τα οποία δεν ανήκουν στην παραδοσιακή κατηγορία των, του καπνού. Είναι μια παγίδα των ε, βιομηχανιών αυτών. Και εγώ καπνίζω, το ξέρετε όλοι, οπότε μπορώ να μιλήσω άνετα, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος καμιανής οργάνωσης κατά του καπνίσματος. Ξέρω όμως πολύ καλά τι προσπαθούν να κάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που θέλουν είναι να συνεχίζουν να κερδίζουν πολλά χρήματα και μάλιστα όλο και περισσότερα χρήματα. Αυτό πρέπει να μπει στην έκθεση, ότι ένα πακέτο τσιγάρων που βγαίνει από το εργαστήριο στοιχίζει 5 σαντίμ. Καταλαβαίνετε τελικά ποιο είναι το κέρδος. Αν το συγκρίνετε με την τιμή πώληση, ακόμα και αν βγάλουμε τους φόρους. Δεύτερον, η καταπολέμηση της απάτης. Γιατί είναι η βιομηχανία του καπνού που τελικά αντιμετωπίζει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απάτη μαζί με την ΟΛΑΦ, ε, είναι αστείο. Είναι σαν να ζητάμε από τον άλλο Καπόνε να δουλέψει για την ε, απαγόρευση του λαθρεμπορίου. Μα δεν έχει καμιά σχέση το ένα με Οπότε δεν είναι δυνατόν να μου λένε, μα μόνο αυτοί μπορούν να ξέρουν κατά πόσο πρόκειται για προϊόντα καπνού που βγαίνουν από μια επιχείρηση ή είναι προϊόντα που έρχονται από αλλού, εγώ το θεωρώ αυτό απαράδεκτο. Η βιομηχανία ε, του καπνού δεν έχει καμιά σχέση με τον έλεγχο αυτό. Πρέπει να εξαιρεθεί. Τρίτον, είναι απαραίτητο, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενισχύσουμε τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει μέσα στους κανόνες αυτούς να ενισχύσουμε και τους κανόνες που έχουμε εδώ στο κοινοβούλιο μας για τους κινδύνους που ελοχεύουν οι συζητήσεις που δεν διέπονται από διαφάνεια με τις διάφορες οργανώσεις. Το 5-3 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο κανόνα. Το έχω πει και πριν από ένα μήνα. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Όλοι έρχονται σε επαφή μαζί σε τον ένα με τον άλλο τρόπο από την βιομηχανία. στη σελίδα σας στο διαδίκτυο, πρέπει να το λέτε αυτό, αλλιώς αντιβαίνετε στους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά έρχομαι στο τελευταίο. Την προηγούμενη εβδομάδα έδειξα με αποδείξεις, έχοντας ε, γράψει κάτι ότι στην ε, υπόθεση Νταλή του Επιτρόπου είχαν πει ψέματα επιχειρήσεις γιατί η σουηδική εταιρεία που ήθελε να επιβάλλει το Σμουθ στην υπόθεση Νταλή είπε ότι είχε συμμετάσχει σε μία συνεδρίαση και από αυτήν κατηγορήθηκε ο Νταλή ενώ δεν είχε λάβει χώρα τέτοια συνεδρίαση και συνέχιζε να λέει ψέματα και αυτό ήταν το κύριο στοιχείο το οποίο οδήγησε στην καθαίρεση του Νταλή, στο να φύγει ο Νταλή. Δεν λέω ότι έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση Νταλή, αλλά είναι σκανδαλώδες να μην έχει πρόσβαση το κοινοβούλιο μας στο φάκελο αυτό. Μόνο οι πρόεδροι και δεν ξέρω καν αν το έχουν δει. Πρέπει να ζητήσουμε διαφάνεια. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση ο Κορεάρ. Μετά Κλάς και μετά Σετζιέσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους μας. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτή την πρόταση οδηγίας. Όπως ελέγχθη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως μια οδηγία που επηρεάζει άμεσα την καλλιέργεια καπνού, αλλά μπορεί να έχει και άμεσο αποτέλεσμα στο παραγωγικό ιστό χωρών όπως είναι η Ιταλία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ισπανία μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους ε, παραγωγούς και την παραγωγή καπνού που είναι κυρίως οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις που δεν χρησιμοποιούν μηχανήματα. Ο κίνδυνος λοιπόν της εξαφάνισης της ε, καπνοπαραγωγή στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα των μέτρων που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν πρόκειται να έχει κανένα αντίκτυπο στην κατανάλωση <clears throat> καπνού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει το 4% του παγκόσμιου καπνού και εισάγει πάνω από 70% του καπνού που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Αλλά το να εξαφανιστούν τα εκτάρια αυτά, τα χιλιάδες εκτάρια που χρησιμοποιούνται στην καπνοκαλλιέργεια θα μπορούσαν, να οδηγήσουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν πολλά κοινωνικονομικά προβλήματα σε περιοχές όπως είναι η Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, όπου περίπου το 25% της αγροτικής παραγωγής είναι καπνοκαλλιέργεια. Επομένως μπορούν να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας που όπως σας είπα αφορούν μικρομεσαίες ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επίσης τα εργατικά χέρια στην επεξεργασία του καπνού και στην καπνοπαραγωγή, στην, συγγνώμη, στην ε, τσιγαροπαραγωγή μπορούν να χαθούν. Η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν δεν είναι σαφές ότι θα αποδειχθεί εις όφελος του Ευρωπαίου καταναλωτή γιατί θα οδηγήσει και σε αύξηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Θα πρέπει να επιδοκιμάσουμε την καλή θέληση της Κομισιόν όταν θέλει να καταστήλει το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, αλλά υπάρχει και μια βασική αντίφαση στην ε, πρόταση αυτή διότι οι προτάσεις τη μπορούν ακριβώς να βοηθήσουν να αναπτυχθεί περισσότερο το λαθρεμπόριο. Σε χώρε όπως η Πολωνία, όπου το 30% της κατανήλωση είναι τα ε, πουράκια με μέντα και στην Βουλγαρία, η απαγόρευση αυτής της κατηγορίας καπνικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη του λαθρεμπορίου για να ικανοποιήσει την παραδοσιακή ζήτηση. Επίση, θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να διαφοροποιήσουμε πλήρω σε αυτή τη συζήτηση την προβληματική της κατανάλωσης καπνού που ξέρουμε όλοι ότι είναι αρνητική για την υγεία και της υποστήριξη για την καπνοκαλλιέργεια. Εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των γεωργών μας και να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση βασίζεται σε στερεά επιστημονικά στοιχεία και εξασφαλίζει την αρχή της αναλογικότητας. Και τέλος, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι αν αυτή η οδηγία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει άμεση επιρροή στις ε, καλλιέργειες, είναι σωστό αυτό το οποίο λέει ο εισηγητής, ότι η Κομισιόν προτείνει να υπάρξουν κατεξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις, τα συστατικά των καπνικών προϊόντων και αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και αβεβαιότητα. Επίσης η Κομισιόν θέλει να έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μειώσει τα όρια νοικοτήνης στα προϊόντα καπνού, κάτι το οποίο μπορεί να έχει και μεγάλη επίπτωση στην πρωτογενή παραγωγή καπνικών προϊόντων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν αν προβλέπει σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επίπεδο να χρησιμοποιήσει αυτή την ε, αυτό το προνόμιο που θέλει και αν θα το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας πραγματικά επιστημονικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Κλάς. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε η κυρία Κορέα σε σχέση με το θέμα της αναλογικότητας. Τι θα πει η αναλογικότητα. Μιλάμε για ένα νομικό, για ένα νόμιμο προϊόν το οποίο βρίσκεται στην αγορά και δεν υπάρχει ένας άλλος τομέας που εμείς να επηρεάζουμε τόσο πολύ προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά. Το ξέρουμε ότι δεν είναι υγιές το να καπνίζει κανείς. Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προσπαθήσει να επηρεάσουμε το κάπνισμα και έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Αλλά το κατά πόσο μια απαγόρευση θα έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό πράγματι το διαμφισβητώ ιδιαίτερα. Οι νέοι ξέρουν, ξέρουμε όλοι ότι ό,τι απαγορεύεται το θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστικό. Σε ό,τι αφορά την προστασία των νέων, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η πρόταση της Κομισιόν για την συσκευασία των τσιγάρων, το λεγόμενο plain packaging, με, μου δημιουργεί το ερώτημα. Είναι πράγματι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίζει πώς θα γίνονται τα, οι συσκευασίες των τσιγάρων. Υπάρχουν κάποιες εταιρείε οι οποίες έχουν ειδικευτεί στα θέματα αυτά και εργάζονται για τις ε, ε, καπνοβιομηχανίες σε σχέση με τον τρόπο, τον βέλτιστο τρόπο να παρουσιάζουν τα πακέτα τους. Γιατί η Κομισιόν θέλει να αναλάβει αυτό το ρόλο και γιατί δεν αφήνουμε αυτό το προνόμιο των εταιριών οι οποίες ξέρουν πώς να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Πώς μπορεί να το αναλάβει αυτό η Κομισιόν και με ποιο τρόπο μπορούν να διαφοροποιούνται τα προϊόντα από μία εταιρεία στην άλλη. Αν εγώ ως καταναλωτής δεν μπορώ να κάνω μια διάκριση μεταξύ των τσιγάρων, άμα δεν ξέρω ποια είναι τα συστατικά τους, άμα έχουν όλα το ίδιο σουλούπι και το ίδιο σχήμα τα πακέτα, πώς μπορώ εγώ να διαλέξω ένα τσιγάρο μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να ξέρω περί πρόκειται. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και θα πρέπει να σκεφτούμε και για το πρόσθετο κόστος το οποίο θα δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό για τον παραγωγό. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ισορροπία και μια αναλογικότητα στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εκπρόσωπη της Κομισιόν αν θεωρεί ότι πράγματι έχει κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν αυτά τα οποία λέει. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο να χαθούν και πάρα πολλέ θέσει εργασία και από τι εταιρείε συσκευασία. Έχει σκεφτεί λοιπόν η Κομισιόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα τη πρότασή τη. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσουν οι πολιτικοί ή γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ένα ενιαίο πακέτο τσιγάρων για όλου του καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Ε, κυρίες και Σιλβέστρης. Ευχαριστώ. Σύντομα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άκουσα τον εισηγητή και πιστεύω ότι είναι πολύ λογικά αυτά τα οποία που λέει. Προσπαθεί να λάβει υπόψη του τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η παραγωγή είναι outsourced, δηλαδή γίνεται από κάποιον εκτός οι αρνητικές επιπτώσεις επίσης θα πάνε εκεί. Θα υπάρχουν, αλλά θα φορούν άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω εσείς πώς θα αναλύσετε την ε, επιρροή που θα έχει η παραγωγή καπνών στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Ίσως θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάει πολύ μακριά, υπερβολικά μακριά. Ευχαριστούμε. Σιλβέστρης και μετά ο κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, και εγώ άκουσα την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θέλει να πετύχει, να κάνει πιο ελκυστικά τα προϊόντα καπνού, να ευνοήσει την εσωτερική αγορά, να το να μειώσουμε το πόσο ελκυστικά είναι τα προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι θα περιορίσουμε και την κατανάλωση. Η πρόταση αυτή Όμως πιστεύω ότι πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή, αν είναι ίδια όλα τα πακέτα, θα εξαφανιστούν διάφορα προϊόντα, τα οποία όμως έχουν κάποιες αγορές σήμερα. Τα slim, για παράδειγμα, τα πιο στενά ε, σιγαρέτα μικρότερης διαμέτρου που είναι με μέντα. Αν υπάρξει τέτοια ομοιογένεια, θα υπάρξει και μια άλλη επίπτωση. Άμα δεν υπάρχουν πια διαφορές ανάμεσα στις μάρκες, η μόνη διαφορά θα είναι η τιμή. Και τι θα μειώσει την τιμή, αν δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα ή κατανάλωση. Είχαμε πει για τον ίνο 30% για, την... για τα σιγαρέτα αυτά θα δούμε τελικά να υπάρχουν περισσότερα παράνομα. Αν δηλαδή ο ανταγωνισμός βασίζεται στην τιμή και μόνο θα πέσει η τιμή. Και θα έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Ο στόχος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία αυτή αντιστρέφονται. Γιατί τελικά ευνοούμε την παράνομη αγορά και έτσι δεν πετυχαίνουμε αυτό το οποίο θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει. Όπως έλεγε πριν και ο εισηγητής ο κύριος Νταβάτζη, η λογική αυτή που λέει ότι οι νέοι καταναλώνουν περισσότερο κάτι το οποίο ξέρουν ότι δεν είναι καλό, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα τσιγάρα που καπνίζω εγώ τι διαβάζω εδώ στο πακέτο. Λένε ότι είναι κακό για την υγεία το κάπνισμα, ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο. Είναι σαφές το μήνυμα. Αν αυτό το γράφουν τα τρία τέταρτα του πακέτου με κάποιες εικόνες πολύ άγριες, ε, δεν νομίζω ότι αυτό θα κάνει την αλλαγή. Ε, αντίθετα, μπορεί οι νέοι να θεωρήσουν ότι είναι cool κάτι τέτοιο και να γίνει της μόδας. Κάποιος ανώριμος νέος, θέλω να πω, όταν έχει να κάνει μια επιλογή, ε, θα προτιμήσει να κάνει κάτι παραβατικό, κάτι που θεωρείται ακριβώς ε, υπερβολικά τολμηρό. Νομίζω δηλαδή ότι με ένα τέτοιο τρόπο μάλλον θα σπρώξουμε τους νέους στην κατανάλωση παρά θα τους απομακρύνουμε. Οπότε με το κείμενό της Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετυχαίνει ακριβώ το αντίθετο από αυτό που θέλει. Δηλαδή θα ενισχύσει την παράνομη αγορά, θα απογορεύσει τα προϊόντα που έχουν μέντα μέσα και επειδή η τιμή τους όπως σας είπα θα μειώσει, θα μειωθεί, τελικά ένας νέος ο οποίος είναι έτοιμος για παραβατική συμπεριφορά θα αρχίσει να καπνίζει αντί για το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πετύχει το αντίθετο αποτέλεσμα πρώτον και δεύτερον κάνει κάτι το οποίο δεν δικιά της δουλειά να είναι ίδια όλα τα πακέτα. Δεν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό, δεν είναι η Ευρώπη που πρέπει να το κάνει αυτό. Αν θέλετε να έχετε μια ενιαία συσκευασία για να μην καπνίζουν οι νέοι, ε, τότε α απαγορεύσουν όλε οι χώρε την πώληση σιγαρέτων σε νέου κάτω των 25. Αυτό θα ήταν πιο λογικό. Αλλά να προσπαθούμε να το πετύχουμε αυτό με τον τρόπο που μας περιγράψανε, πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικό και ότι το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Τέλος. Τέλος. Διαβάζω εδώ πάνω στο πακέτο τσιγάρων ότι είναι αρνητικές οι επιπτώσεις από το κάπνισμα και για σας και για τον περίγυρό σας. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν οι νέοι να βρίσκουν εύκολα τσιγάρα και να μην μπορούν τόσο εύκολα να έχουν πρόσβαση στα τσιγάρα. Είναι άλλο για τον περίγυρό μας. Αυτό η οδηγία δεν το τρει. Υπάρχουν αεροδρόμια, μάλλον δεν τηρεί την ελευθερία να μπορεί κάποιο ο οποίο επιλέγει να καπνίσει να το κάνει. Ορισμένα αεροδρόμια δεν έχουν τέτοιο χώρο όπου να μπορούν να πηγαίνουν οι καπνιστές και να καπνίζουν. Οπότε τελικά τι κάνουν οι άνθρωποι, ε, μπορεί να πάνε στις τουαλέτες να καπνίσουν, άμα δεν έχουν κάτι άλλο. Και αυτό είναι κακό φυσικά για τον περιγυρό μας. Πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα των καπνιζόντων, άμα δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στους δικούς μας, σε αυτούς που είναι γύρω μας. Και οι φωτογραφίες αυτές που λένε για τον καρκίνο του πνεύμονα, και ότι το κάπνισμα δημιουργεί αυτό τον καρκίνο να βάλουμε και τη γιαγιά μου, η οποία πέθανε 92 ετών και κάπνισε μέχρι την τελευταία μέρα. Να βάλουμε και αυτή τη φωτογραφία τότε, δίπλα σε αυτές που προτείνεται των πνευμόνων των καπνιστών. Ναι, μπορούμε από τη μια μεριά να βάλουμε το ένα, από την άλλη μεριά θέλω Να σας δώσω τη φωτογραφία της γιαγιάς μου, άμα θέλετε, και με τη βεβαίωση ότι παρόλο που κάπνιζε δύο πακέτα την ημέρα, έζησε μέχρι τα 92 της. Ε, προφανώς η, η προάσπιση της δημόσιας υγείας είναι μείζον υποχρέωση όλων μας. Εδώ όμως δεν μιλάμε για την απαγόρευση των προϊόντων καπνού, μιλάμε για τη ρύθμιση της αγοράς τους. Και αυτό για το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την Επιτροπή μας είναι ότι θα πρέπει με σαφήνεια να γίνεται διάκριση μεταξύ των προσμίκτων των αρωματικών που κάνουν πιθανώς ελκυστικότερα στους νέους τα ε, προϊόντα του καπνού με εκείνα τα πρόσμητα τα οποία είναι απαραίτητα για να είναι αξιοποιήσιμα και άρα εμπορεύσιμα τα ευρωπαϊκά καπνά στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Τα, τα καπνά δηλαδή Μπέρλεϊ και ανατολικού τύπου. Και δεν πρέπει να διαφεύγει της Επιτροπής μας ότι εάν δεν γίνει αυτή η διάκριση τότε μιλάμε μοιραία για την απομάκρυνση από την αγορά των ευρωπαϊκών καπνών, τη θέση όμως των οποίων θα πάρουν τα καπνά, τα Βιρτζίνια που έρχονται από τις τρίτες χώρες. Αυτό είναι και αφελές και καταστροφικό βεβαίως για τους 500.000 Ευρωπαίους παραγωγούς καπνών, οι οποίοι δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι αποτελούν κυρίως μέρη του αγροτικού πληθυσμού που βρίσκονται σε περιοχές με πάρα πολλούς περιορισμούς. Είναι συνήθως μονοκαλλιέργεια τα καπνά για τους ανθρώπους αυτούς και το κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί θα είναι τεράστιο. Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ είναι η, πρόταση για, την, ε, για τη μη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ε, τσιγάρων, η, η ενιαία δηλαδή σήμανση δεν, ε, δεν έχω καταλάβει ε, πώς η Επιτροπή νομίζει ότι αυτό το μέτρο θα είναι αποτελεσματικό. Αυτό όμως που πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που θεωρώ ότι μια τέτοια αντιμετώπιση ε, δημιουργεί είναι ότι αποστερούμε από τις βιομηχανίες καπνών να έχουν οποιοδήποτε λόγο, οποιοδήποτε κίνητρο να βελτιώσουν την ποιότητα των δικών τους προϊόντων και να τα κάνουν λιγότερο βλαβερά προς τους καταναλωτές. Τέλος, θέλω μία ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Με ποια λογική, με ποια επιχειρήματα και μετά από ποια μελέτη θεωρείτε ότι η απαγόρευση που θεωρώ ότι είναι αυθαίρετη απόλυτα της παραγωγής των, των τσιγάρων slim θα είναι θετική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Σας ευχαριστώ Σπύρο. Τελείωσαν τώρα οι παρεμβάσεις. Λίγα λεπτά μόνο στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, στην κυρία Γουέλμερ. Μετά εσεί να απαντήσετε κύριε Ταμπάζνη. Ορίστε παρακαλώ κυρία μου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες από τις απαντήσεις ελπίζω έγινε μία αναφορά σε όρια ηλικίας και ότι ιδεοδός θα έπρεπε η οδηγία να προβλέπει και ηλικίες. Ωστόσο, η νομική βάση του 114 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει στην Ένωση να βάλει ως βάση ε, σε νομοθεσία όρια ηλικίας. Έγιναν τώρα διάφορες παρεμβάσεις σχετικά με την διαφοροποίηση μεταξύ προϊόντων και προτάθηκε ε, μάλλον ε, ισχυρίστηκε κάποιο ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι δυνατό. Εμεί δεν νομίζουμε να συμβαίνει αυτό. Πρώτα, για να διευκρινίσουμε, η πρόταση τη Κομισιόν δεν αναφέρεται στο plain packaging, ούτε στην κατάργηση όλων των συστατικών γεύσης στα προϊόντα καπνού. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος, επαρκές περιθώριο για τις ε, εταιρείες καπνού ώστε να μπορούν να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους στην αγορά και οι καταναλωτές επομένως να μπορούν να επιλέγουν και όχι μόνο στη βάση της τιμής. Σε ό,τι αφορά την αφαίρεση των επιπέδων TNCO, αυτά τα έχουμε δει σε πολλά επιστημονικά φόρα τον τελευταίο καιρό. Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι αν αγοράσουν ένα πακέτο που να μην έχει 10 χιλιοστόγραμμα πίσας αλλά μόνο 8 ότι κάνουν κάτι καλό για την υγεία τους. Γι' αυτό οι επιστήμονες σήμερα προτείνουν αντικατάσταση αυτών των ενδείξεων TNCO με ποιοτικέ προειδοποίησεις και αυτό προβλέπει η πρόταση Κομισιόν. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες αναφέρθηκαν πλήρωνες ευρωβουλευτές. Οι πράξεις που προτείνονται στην πρόταση οδηγίας προβλέπουν συγκεκριμένες ενδείξεις που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή, από την Κομισιόν δηλαδή, και θα επιτρέψουν την συμπερίληψη νέων επιστημονικών δεδομένων. Και εδώ συμφωνούμε με τους βουλευτές οι οποίοι αναφέρθηκαν, παρέπεμψαν στα επιστημονικά δεδομένα. Θεωρούμε και εμείς ότι ό,τι γίνεται στο επίπεδο της Ένωσης πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα και καλύτερα επιστημονικά δεδομένα. Γι' αυτό, για να μπορέσει να περιλάβει η Κομισιόν τις επιστημονικές εξελίξεις, χρειαζόμαστε έναν αριθμό από κατεξουσιδότηση πράξης. Για τον υπολογισμό σχετικά με την επίπτωση στην απασχόληση, ναι βέβαια αυτό ήταν σημαντικός παράγον στην μελέτη επιπτώσεων και βεβαίως ο καθένας μπορεί να εξετάσει το έγγραφο. Με δύο λόγια, εμείς καταλήξαμε με τους υπολογισμούς μας ότι η εφαρμογή της προτάσεως μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 5.000 θέσεων εργασίας στα 5 χρόνια μέσα στην Ένωση, που όμως θα αντικατασταθούν από 8.000 άλλες θέσεις εργασίας σε όλη την Ένωση μέσα στην πενταετία. Είδαμε και εξετάσαμε δηλαδή τις βιομηχανίες και στα ανάντι και στα κατάντι της καπνοβιομηχανίας. Τώρα για τα σιγαρέτα Slim. Απαγορεύονται στην πρόταση διότι έχουν παραπλανητικό αποτέλεσμα. Εάν εξετάσετε τα νούμερα των πωλήσεων σιγαρέτων Slim την τελευταία πενταετία, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκαν οι πωλήσει τους κατά 50% μέσα σε ένα συνολικό σενάριο μείωση της κατανάλωσης. Άρα η αύξησή τους είναι δυσανάλογη στην Ευρώπη και αυτό εν μέρη οφείλεται στο γεγονός ότι παραπλανώνται οι καταναλωτές επειδή θεωρούν ότι είναι λιγότερο επιβλαβή για την υγεία τους. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Γενική Διεύθυνση Σάνκο. Συνοψίζει ο κύριος Τσάμπα Ταμπάζδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα γιατί να μην ζητήσουμε και τη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, γιατί δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα για τη μελέτη επιπτώσεων για, στους γεωργούς, στους αγρότες δηλαδή, ποια θα είναι, ποιες θα οι επιπτώσεις της οδηγίας αυτής στους αγρότες. Εγώ δεν έχω δει τέτοια μελέτη επιπτώσεων και όμως ε, ασχολούμαι το θέμα αρκετό καιρό. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ας ακούσουμε και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και ας επανέλθουμε να ρωτήσουμε και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν απήντησε στην ερώτηση. Όταν είπε ότι θα χαθούν 5.000 θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής εμείς δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η επίπτωση στους αγρότες. Δεν μας έχουν δοθεί συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε για το παράνομο εμπόριο. Για το πώς προτίθενται να μειώσουν το παράνομο εμπόριο. Συμφωνώ με την κυρία Κλάς και άλλους συναδέλφους που είπαν ότι το σκέτο πακέτο, το plain packaging, γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας και είναι κέριο πρόβλημα για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Κάποιος συνάδελφος είπε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να λέει επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα και εξαιρετικά επικίνδυνα. Αυτό είναι απλός τρόπος για να επικοινωνήσει κανείς με τους καταναλωτές και να τους κάνει να αντιληφθούν πόσο επικίνδυνα είναι τα προϊόντα. Ο Σπύρος αλλά και άλλοι συναδελφοί μου είπαν ότι πώς θα επιλέξουν οι καταναλωτές μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. Γιατί βέβαια όλα τα προϊόντα καπνού είναι, ε, είναι βλαβερά, αλλά όχι το ίδιο. Δεν είναι όλα το ίδιο βλαβερά. υπό την ισχύουσα νομοθεσία δεν δίνεται απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι βέβαια πρόβλημα υγείας και γι' αυτό είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΚΟ. Για την προστασία τώρα των καταναλωτών πρέπει να επανεξετάσουμε ολόκληρο το θέμα της αξιόπιστης ενημέρωσης. Συμφωνεί η Επιτροπή Γεωργίας ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ παραγωγών και βιομηχανιών του καπνού. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μποβέ ότι η μεγάλη καπνοβιομηχανία δεν έχει καμιά αναστολή. Δεν την απασχολούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Στην οδηγία αυτή μεταξύ άλλων μέτρων, θα πρέπει να επιβάλλουμε πλήρη απαγόρευση σε οποιαδήποτε άλλα παρόμοια προϊόντα. Για παράδειγμα, αυτά τα τσιγάρα, αυτή, μάλλον αυτές τις τσίκλες που μοιάζουν με τσιγάρα, πρέπει να απαγορευτούν αυτά τα πράγματα. Τα οποία προσελκύουν σιγά σιγά τα μικρά παιδιά στο, στην ιδέα του καπνίσματος. Να, έχετε αυτές τις τσίκλες που μοιάζουν με τσιγάρα. Αυτά δεν είναι δυνατόν να τα ανεχθούμε. Θα δώσω τελική μορφή στην οδηγία, στην πρότασή μου δηλαδή, τις επόμενες εβδομάδες και θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Εντάξει αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνει εδώ η συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 24-25 Απριλίου. Για αυτούς που δεν θα δω, καλό Πάσχα. Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα γίνει η συνεδρία των συνατονιστών. Οι και οι συγητές ακολουθούν. Σε δύο λεπτά.